Okay, dear colleagues, I would like to start our meeting. Να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω όλους. Να κάνουμε δεκτή πρώτα την μέρησια διάταξη. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες... Um, on you know, the agreement, since no amendments για τη συμφωνία με την Νορβηγία για το ΦΠΑ δεν έχουν υπογραφεί, δεν έχουν κατατεθεί τροπολογία στην έκθεση του Μιγγέλ Βιέγα για τη συμφωνία με την Νορβηγία για τον ΦΠΑ, οπότε δεν θα γίνει συζήτηση επί των τροπολογιών και θα περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία τη έκθεση αύριο στι 24 Απριλίου. Οι συστάσει και αποφάσεις μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών της 26 Μαρτίου το επόμενο θέμα. Έχουμε καταρχάς εκθέσει πρωτοβουλίας σειρά προτεραιότητας ε, των εκθέσεων δύο πρωτοβουλίας από την ΕΚΟΝ και για την ποσόστοση έχουμε την αιτήσια έκθεση για τη ΣΥΜΠΗ, την ΕΚΤΑ για την αιτήσια έκθεση τον ανταγωνισμό και αιτήσια έκθεση για την ΕΤΕΠ. Επίσης θα ζητηθεί παρέκκληση από τι αποφάσει τη Πολιτική Ψηφοδέλφου 15η Μαρτίου, ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε εξοδότηση για να προετοιμάσουμε για τα τρία αυτά θέματα και επίσης εκτός ποσόστοσης ετήσια έκδοση για τραπεζική ένωση. Το επόμενο, για τα επόμενα βήματα στις διαδικασίες διορισμού ε, της ΕΚΤ συμφωνήσαν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για το διάλογο με Συμβούλιο Eurogroup σε σχέση με αναβασμένο ρόλο του Κοινοβουλίου, για τις ε, ε, διορισμούς, ιδίως αυτών που θα διαδεχθεί τον ε, διοικητή της ΕΚ. Για τον Brexit τώρα συμφωνήσαμε για τα περαιτέρω στοιχεία της μεθόδου εργασίας και υπάρχει και αύριο μία συνάντηση στο πλαίσιο και τις έκθεση σχέσεις που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί οι συντονιστές συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ευθυγράμμιση και συνέπεια στο Κοινοβούλιο μεταξύ των θέσεων της Επιτροπής τελευταίος ε, πάλι Ernst και ε, Η γραμματεία θα μεταφράσει κάποιες πληροφορίες για τις δημοσιακροάσεις. Ε, ακρόαση για το ΦΠΑ. 24 Απριλίου εγκρίθηκε το σχέδιο προγράμματος με προσθήκες. Σε σχέση με κάποια προβλήματα με την πώληση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων θα έχουμε μία ειδική συνάντηση με το θεματικό τμήμα. 19 Ιουνίου έχουμε εμπειρογνώμονε. Γαλλία, Ιταλία, NCA, ένα εκπρόσωπο από τι Ευρωπαϊκέ Εποπτικέ Αρχέ ΕΙΟΠΑ, ένα εκπρόσωπο από την Επιτροπή και έναν εκπρόσωπο από το Better Finance. Επίσκεψη αντιπροσωπεία για την επίσκεψη εβδομάδα Βασιλείας ε, δεν έχουμε σχόλια. Και σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ θα περιληφθεί η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον. Οικονομική διακυβέρνηση. Θα ζητήσουμε ευκολίες για να έχουμε μια έκτακτη συνάντηση 9 Ιουλίου Δευτέρα, 3 το μεσημέρι για το νομισματικό διάλογο και την ακρόαση SRB. Μάριο Ντράγκη θα είναι πάρουν και στα δύο αυτά. Οι συντονιστές συμφώνησαν περαιτέρω στοιχεία τη συνέχεια που θα δοθεί στο πακέτο του Δεκεμβρίου για την ΟΝΕ και συμφώνησαν να προσκληθούν ορισμένα μέλη του ε, Εποπτικού Συμβουλίου του Μηχανισμού Εποπτείας σε μία συνάντηση και κλεισμένο τον θεωρώ αύριο θα υπάρχουν κάποιοι επόπτες ε, από, την, από το Ευρωπαϊκό Εποπτικό Συμβούλιο που θα παρέ, παρίστανται. Σε ό,τι αφορά πιθανές μελικές μελέτες από το θεματικό τμήμα, επειδή κοντεύει να λήξει θητεία, φάση συντονιστέ, μόνο μία μελέτη να γίνει σε σχέση με τον αντίκτυπο του κανονισμού 537 του 2014 για κόστος, συγκέντρωση, ανταγωνισμό στην αγορά καταστατικών ελέγχων. Για τι αναφορές δεν χρειάζεται να δοθεί συνέχεια στι αναφορές. 56 του 17 και 429 του 17. Προτάσει ψηφίσματος. Δεν θα δοθεί συνέχεια στην πρόταση ψηφίσματος Β8. 131 κάθετος 2018 για την ε, συνεργατική οικονομία. Επίσης, ε, αίτηση έκθεση πρωτοβουλία στην Επιτροπή Γυναικών. Θα ζητήσουμε κανόνα 55 να βγει δηλαδή το σλότ μόνο από την Επιτροπή ΦΑΜ. Αλλιώ δεν το δεχόμαστε. Μόνο κανόνα 55. Και δεν είχαμε κάποια άλλη αντίρρηση για τα σχολονοθυρίδε ε, και τι συναντήσει ε, με την Οικονομική Επιτροπή τη Μπούντε τα 19 Ιουνίου και την Κοινή Επιτροπή με την ΕΜΠΛ για τι ειδικέ τάσει αναχώρα 28 Ιουνίου. Για το πρότυπο χρηματοπιστικής πληροφόρηση 17, στα διάφορα συμφωνήθηκε να κατατεθεί πρόταση ψηφίσματος για την Ολομέλεια του Ιουλίου στο 3. Τώρα να σας πω τι γίνεται με τους τριμερείς διαλόγους. Ε, το τριμερή διάλογο για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 10 Απριλίου. Καταφέραμε τα τρία θεσμικά όργανα να καταλήξουμε σε προσωρινή συμφωνία. Θα υπάρξει εκ νέου διαπλήσεων την Επιτροπή με βάση το κανόνα 69F του κανονισμού. Περιμένουμε βέβαια την επίσημη βεβαίωση της έγκρισης της συμφωνίας από το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το οργανισμό ECN-SIN, 17 Απριλίου, είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν με το χρονοδιαγράμματος, και πώς θα συζητηθούν τα πολιτικά και τεχνικά άρθρα. Χωρίστηκαν δηλαδή κάποια άρθρα σε πολιτικά και κάποια άλλα σε τεχνικά. Υπάρχουν κάποια ζητήματα όπως ε, η ανεξαρτησία, οι πόροι, τα πρόστιμα, οι κατασφαλιστές και τα λοιπά που άνοιξαν χωρίς κατάληξη, να καταλήξουμε συμφωνία. Θα έχουμε επόμενο τριμερή διάλογο 14 Μαΐου, 30 Μαΐου και προπαρασκευαστικό έργο σε τεχνικό επίπεδο στο μεταξύ. Τέταρτο, έγκριση των πρακτικών της συνάντησης 19-20 Μαρτίου, 26-27 Μαρτίου, 9 Απριλίου, όλα του 18, αν δεν υπάρχουν σχόλια. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Και επιτέλους μπορούμε να πάμε στο σημείο 5 που είναι η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά ε, τη ρύθμιση και την εποπτεία χρηματοπιστικών υπηρεσιών. Brian Hayes είναι ο εισηγητής. Θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης του συγγητού αφού μας κάνει μια αποκαταρκτική παρουσίαση. Έχετε το λόγο κύριε Χέις; Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία η έκθεση αυτή για δύο λόγους. Πρώτον, τον προηγούμενο Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν κατάλογο στον τομέα των, των χρηματοπιστωτικών των αποφάσεων περί ισοτιμίας. και μετά έρχεται το Brexit, κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ανεξάρτητα τη γνώμη που έχουμε για το Brexit θα πρέπει να υπάρξει μια εκ νέου ευθυγράμμιση ανάμεσα στις θέσεις μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και τις θέσεις της διαπραγμάτευσης που θα συζητηθούν στη διαπραγμάτευση ή που συζητιούνται ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. <clears throat> Βασικός στόχος λοιπόν της έκθεσης αυτής είναι να προσπαθήσει να κάνει μια επιβλέψη αν θέλετε ο οριζοντίου τύπου των αποφάσεων ισοτιμίας. Καταρχάς να δούμε αν είναι χρήσιμες οι διαδικασίες αυτές, είναι βελτιώσιμες. Μπορεί το σύστημα των ισοτιμιών να είναι πιο υπόλογο σε έλεγχο και βλέποντας τις αποφάσεις είναι σαφές ότι το υπάρχον πλαίσιο ισοτιμιών ως έχει είναι σαφές ότι χρειάζεται πολλές βελτιώσεις. Δεν έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για τις ισοτιμίες, λαμβάνονται κατά περίπτωση οι αποφάσεις και διαφέρουν για κάθε θέμα. Μία από τις συστάσεις μου είναι να υπάρχει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση ισοτιμιών. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία τυποποιημένη διαδικασία για τη λήψη των αποφάσεων ισοτιμιών. Το ενιαίο πλαίσιο αυτό θα διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη συνεκτικότητα και στον τρόπο λήψης αποφάσεων αναφάκελων. Θα πρέπει επίσης να πούμε στα πλαίσια της σωστής και πλήρους εξέτασης του θέματος αυτού από το Κοινοβούλιο αν η ισοτιμία είναι το καλύτερο μέσο για να ασχοληθούμε με τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Μια απόφαση για ισοτιμία είναι μια μονομερής απόφαση που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χορηγήσει σε όργανα τρίτων χωρών πρόσβαση στις αγορές μας. Είναι θα έλεγα μονόδρομη επικοινωνία, δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν μήπως θα πρέπει να προσβλέπουμε σε ένα σύστημα πληρέστερο αμοιβαίας αναγνώρισης και αμοιβαίας πρόσβασης και όχι σε μονομερείς αποφάσεις. Σίγουρα κάτι τέτοιο θα είναι πιο δύσκολο. Από την άλλη όμως θα έχει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα για τα οικονομικά όργανα, τα χρηματοπιστωτικά όργανα και την πρόσβασή τους σε τρίτες αγορές. Παραδέχομαι ότι οι ισοτιμίες δεν ή μάλλον ευνοούν εν πολλής την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως η καταγραφή των επιχειρήσεων, η ποικιλία των προγραμμάτων, των προϊόντων, οι κεφαλαιοκικές ροές και η επιβολή των διεθνών επιπέδων τυποποίησης και της μείωσης των συστημικών κινδύνων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο όμως δεν κρύβει τους κινδύνους που υπάρχουν και εφαρμόζονται με ακριβώς εφαρμοστικές πράξεις. Το Κοινοβούλιο δεν έχει εδώ τίποτα να παίξει σαν ρόλο. Οι αποφάσεις μας είναι τεχνικής φύσεως και όχι τόσο πολιτικής φύσεως. Στην έκθεσή μου αναφέρομαι στην απόφαση για την Ελβετία του Δεκεμβρίου του 2017 η απόφαση αυτή ε, είναι περιορισμένη χρονικά, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα εξαρτηθεί η παράτασή της από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο. Εγώ δεν λέω αν ήταν σωστός αυτός τρόπος. Το θέμα είναι αν η απόφαση αυτή είναι πολιτική απόφαση και αν ναι, γιατί το Κοινοβούλιο δεν έχει ουδεμία εμπλοκή. Όπως είπα και στην έκθεση Μπάλτς, για τον κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κανονικά οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται μάλλον μέσω μιας κατεξουσιοδότησης πράξης. Είναι συνεπώς ε, ένα σημαντικά, σημαντικά πολιτικό ε, ε, περιεχόμενο και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συνυπογράφει τις συμφωνίες και να παίζει έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για τις ισοτιμίες. Κάνουμε και κάποιες προτάσεις για την τακτοποίηση της διαδικασίας ε, για τις ισοτιμίες. Είπαμε ότι θα πρέπει να ανανεώνονται ανά από την αρμόδια αρχή. Η εποπτεία θα πρέπει να διεξάγεται επίσης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές έτσι ώστε οι τρίτες χώρες ε, να σέβονται τους κανόνες και επίσης προτείνουμε να υπάρξουν πιο ξεκάθαρες διαδικασίες για την υιοθέτηση, κατάργηση και αναβολή εφαρμογής μιας αποφάσεως ισοτιμίας. Και θα πρέπει να δούμε επίσης πώς θα συνεργαστούμε και με τα διεθνή διαιτητικά σώματα σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη που υπάρχει για μια διεθνώς πιο συνεκτική αντιμετώπιση των δημοσιονομικών θεμάτων έτσι ώστε να βελτιώσουμε την διεθνή ισορροπία και τις ανισότητες. Συνεπώς λοιπόν εγώ προτείνω κάποιες ιδέες για το πώς θα συνεχίσουμε σε σχέση με τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, σε σχέση με το Brexit και περιμένω από τους σκιώδεις και τους συναδέλφους έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε καταλήξει σε μια κοινή προσπάθεια καθοριστική του μέλλοντός μας στον τομέα της χορήγησης ισοτιμιών. Ευχαριστώ. Χουάν Φερνάντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, μια πάρα πολύ απαραίτητη όπως είπε και ο εισηγητής έκθεση. Αλλά είναι, δεν είναι δυνατόν μάλλον να αποσυνδέσουμε τη συζήτηση για την έκθεση αυτή από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, ε, ιδιαίτερα το θέμα της, ε, <clears throat> του Brexit σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πιο τεχνική και λιγότερο πολιτική συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία να έχει σαν στόχο τον εναρμονισμό των διαφόρων ισοτιμιών και να προσπαθήσουμε να ορίσουμε σωστότερα τα κριτήρια για τα συστήματα ισοτιμίας που υιοθετούμε κάθε φορά σε κάθε κανονισμό και σε κάθε νομοθετική πράξη και οδηγία. Συνεπώς λοιπόν <clears throat> βλέπουμε ότι ε, έχει γίνει πρωταγωνιστής της θέματο, του θέματος αυτού το Brexit. Πέρα από τα τεχνικά θέματα τίθεται γενικά το πρόβλημα του πώς θα λειτουργήσουν τα συστήματα ισοτιμίας στο μέλλον. Δεν πρέπει λοιπόν να αποκρύψουμε την σημασία της έκθεσης αυτής σε μια τόσο κομβική στιγμή και θα πρέπει να διευκολύνουμε το Κοινοβούλιο να υποδείξει κάποιες ε, κατευθύνσεις για τους διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιου είδους θέματα. Είναι σημαντική η έκθεση αυτή, είναι επαρκής, είναι εύθετη χρονικά Νομίζω η δουλειά την οποία μας έχει προτείνει μέχρι τώρα ο εισηγητής είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θέλω να τον ευχαριστήσω, να τον αναγνωρίσω γιατί καταγράφει μια σειρά αρχών και μια σειρά αξιών επί των οποίων θα μπορέσουμε να διαιτητεύσουμε του συστήματος των νοσοτιμιών και να μπορέσουμε σαν κοινοβούλιο να πρωταγωνιστήσουμε, να ενισχύσουμε τον ρόλο μας, να γίνουμε πιο σημαντικοί, ιδιαίτερα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα <clears throat> δεν είναι εύκολα. Δεν είναι ε, ξεκάθαρα μερικές φορές ε, ε, ποιοι είναι οι στόχοι του εισηγητή, γι' αυτό και θα καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες τις επόμενες εβδομάδες. Το σύστημα χορήγησης ισοτιμίων είναι κεντρική σημασίας. Στόχος είναι η αμοιβαία αναγνώριση ε, που προτείνεται στην παράγραφο 5 δεν έχει την σωστή διατύπωση. Νομίζω ότι επίσης και στην παράγραφο 8 οι προτάσεις ε, για τις ισοτιμίες εντάσσονται γενικότερα στο πλαίσιο των νομοθετικών εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι γενικότερα σε επίπεδο διεθνών συμφωνιών λαμβάνονται υπόψη ακριβώς και το τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές, αλλά για να μην υπάρχουν μόνο ξεκάθαρα, το λέμε, ε, αμοιβέ αναγνωρίσεις, θα πρέπει να δούμε τι ισχύει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με το 17, στο 17 δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ενός αυτόματου συστήματος χορήγησης ισοτιμιών, ακούγοντας τον εισηγητή δεν είναι ξεκάθαρο το πώς ε, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε δυνατότητες αύξησης του ρόλου του Κοινοβουλίου σε πολιτικό επίπεδο, αλλά έτσι όπως περιγράφεται στο 17 και στο 19, ε, οι εποπτικές αρχές, η ΕΣΜΑ, η ΕΙΟΠΑ, η EBA, δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος και νομίζω ότι η κατάσταση σίγουρα και στο άρθρο 20 σχετικά με τις εθνικές εποπτικές αρχές νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε να στηρίξουμε κάποιες από τις προτάσεις που περιλαμβάνει το 20. Πάντως είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε την συζήτηση αυτή είναι σαφές ότι η έκθεση αυτή δεν μπορεί να αποκολληθεί από τη συζήτηση για το Brexit. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις συνέπειες του Brexit στα πλαίσια της συζήτησης συγκεκριμένης έκθεσης. Δεν θα μείνουμε μόνο σε τυπολογικού τύπου παρατηρήσεις αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική για όλους συμφωνία έτσι ώστε η Ευρώπη να έχει ένα σύστημα ισοτιμιών αμοιβαία αναγνωρίσιμες αν είναι δυνατό να γίνει αυτό αλλά οικονομικά συμφέρουσες που να καλύπτουν και τη νέα πραγματικότητα του Brexit. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάτσεκ από τους Φιλελεύθερους, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο εκθεσής του. Τονίζει σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη, όχι μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με το μεγαλύτερο τμήμα της, των προτάσεων του εισηγητή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει και θα εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις με τις τρίτες χώρες όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε διαπραγματεύσεις ε, για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του μεγαλύτερου κέντρου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Υπήρου μας. Επίσης, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος ε, έχει την πρόθεση να ανακαλέσει ε, όλες τις, όλες, ό, όλους τους τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης ε, που υπήρξαν μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να έχουμε συναλλαγές ε, με τις τρίτες χώρες ε, που δεν είναι στη δικαιοδοσία μας. Υπάρχουν πολλά ωφέλη όσον αφορά τις διατάξεις οδυναμίας, για παράδειγμα διευκόλυνση των συναλλαγών σε διασυνοριακό επίπεδο, υψηλά πρότυπα εποπτείας, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονό ότι είμαστε η μοναδική δικαιοδοσία στον κόσμο που δίνει τη δυνατότητα ισοδυναμίας ε, στο δικό τη σύστημα. Δεν είναι εντελώς ολιστική η προσέγγιση μας, είναι κατά περίπτωση ανανομοθεσία δηλαδή. Και σε έναν ιδανικό κόσμο θα έπρεπε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε πιο συνεκτικές ε, διαδικασίες ισοδυναμίας ε, με μεγαλύτερη ε, δημοκρατική λογοδοσία που δεν θα βασίζονται μόνο σε πολιτικά κριτήρια. Βέβαια είναι αβέβαιο το τοπίο και πρέπει να διατηρήσουμε τα υψηλά μας πρότυπα αλλά θα διατηρήσουμε και μια ανοιχτή αγορά. Η συνεργασία συνεργασία με τις, χώρες, με τις τρίτες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι Ένα αρμονισμένο πλαίσιο εξασφαλίζει ότι διατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο τα πρότυπα. Όμως ε, όταν ε, θέλουμε να καλέσουμε τρίτες χώρες να προβούν σε συναλλαγές στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους ε, ρυθμιστές, με τις ρυθμιστικές αρχές των χωρών αυτών, ε, να μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε αυτήν την ήπια δύναμή μας ε, σε διεθνή φόρα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ευθυγράμμιση ρυθμιστική και εποπτείας. Με τα εργαλεία λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο Φίλιπ Λάμπερτς. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Δεν ενημερώθηκα και για να μην σπαταλήσω το χρόνο σας, καλύτερα γραπτός να υποβάλω τις παρατηρήσεις μου, αντί να πω ανοησίες ε, επειδή κάποιο μου είπε ότι είπα νοησίε την περασμένη μου εβδομάδα στην Ολομέλεια, με έχει πιάσει μια συστολή. Δεν θα πω τίποτα λοιπόν. Δεν βλέπω κανένα από την Google, λέει ο πρόεδρο. Η FDD. You are speaking for the FDD. Μιλάτε εκ μέρου του FDD. Ε, ε, ελπίζω. Ελπίζω. δεν πρέπει να κάνετε διακρίσεις κατά της Μεγάλης Βρετανίας και κατά του City. Ε, πρέπει να πριτανεύσει η λογική ως προς αυτό. Υπάρχουν όμως πολλές προκαταλήψεις γιατί εμείς ασκούμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δικαίωμά μας. Εσείς ε, θα έπρεπε να θέλετε να συναλλάσσεστε μαζί μας όμως γιατί εμείς είμαστε οι τραπεζίτες της Ευρώπης στο Λονδίνο και δεν θα θέλατε να κάνετε κάτι που να είναι εναντίον μας. Ε, γι' αυτό προτείνω να το λάβετε και αυτό υπόψη. Το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι. Thank you. Ευχαριστώ. ENF, sorry. We have... ENF, έχουμε κανένα από την ENF. Όχι. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στο Catch the Eye. Yes, Vance Perez. Merci, Monsieur. Vance Perez. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Με την έκθεση αυτή πρωτοβουλίας ε, η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή μας μπαίνει στην, ουσία της ε, συζήτηση και στο δύσκολο κομμάτι της συζήτηση ε, για την ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ε, είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μετά από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Φεβρουάριο του 2017 και είχε γίνει μια ανταλλαγή απόψεων τότε με τον Γενικό ε, Διευθυντή της ΦΙΣΜΑ ε, για αυτό το καθεστώς ισοδυναμίας. Εγώ με ένα πράγμα ε, συμφωνώ ε, σε αυτά που είπε ο εισηγητής, ότι το καθεστώς ε, ισοδυναμίας όπως υπάρχει, όπως εξακολουθεί να υφίσταται μετά μέσα από αυτό το ιδιαίτερο, με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να προσαρμοστεί λόγω της επερχόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως μου φαίνεται ότι πέρα από αυτό ε, βλέπουμε διαμετρικά αντίθετα ε, το όλο ε, θέμα. Ενδεχομένως το καθεστώς ισοδυναμίας να μην είναι κατάλληλο για το σκοπό που προσπαθεί να επιτύχει. Αλλά μπορούμε να πούμε δύο διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτό. Ο εισηγητής προτείνει προφανώς απλώς να ε, ένα σύστημα το οποίο ε, έχει δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα επίπεδο απαιτήσεων ε, πολύ υψηλό όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία οντοτήτων τρίτων χωρών σε ένα πλαίσιο ενιαίας αγοράς σε πνεύμα πολύ ανοιχτό και αυτό προς που είναι κατεστημένες σε τρίτες χώρες αλλά δεν καταλαβαίνω καταλαβαίνω ε, αυτό το κατάλληλο για το σκοπό που θέλει να επιτύχει ε, που είπε ο εισηγητή στο πλαίσιο του καθεστώτο ισοδυναμία και επενθυμίζω ότι αυτό είχαμε πει ότι είναι το σωστό καθεστώ ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που, γίνεται, που γίνονται αυτή τη στιγμή από τον Μισελ Μπαρνιέ. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά από τον εισηγητή, θέλει να περάσουμε σε ένα καθεστώ αμοιβαία αναγνώριση με αυτό θέλει να ανταλλάξει το τρέχον σύστημα. Υπάρχει ένας κίνδυνος όμως που αναλαμβάνουμε. Ο εισηγητής μας προτείνει όχι να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα είναι το καλό παράδειγμα ε, να μην υπάρχει δηλαδή μια πρόταση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το θέμα αυτό, αλλά να αποδυναμώσουμε κάπως και να προσαρμόσουμε ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία στη διεθνή νομοθεσία, στις ανάγκες της διεθνής νομοθεσίας. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία, τη γνωρίζουμε πολύ ε, και εδώ τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Ε, δεδομένη της χώρας από, τις, ε, από, την οποία προέρχεται ε, πρέπει να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί είναι ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τη χώρα αυτή όμως δεν είναι η μόνη χώρα για την οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αντίκτυπος αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή νομοθεσία και εγώ πιστεύω γι' αυτό ότι πρέπει οπωσδήποτε να βασιστούμε στην προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να, βασιστήσουμε, να βασιστούμε στην ε, θέλησή μας να καταλήξουμε σε μια διαδικασία ισότιμης μεταχείρισης, κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, δεν θα βρίσκονται ε, πλέον σε μειονεκτική ε, θέση, δεν θα χάσουν λόγω αυτής της νέας διαδικασίας και να λαμβάνονται υπόψη και τα ωφέλη των ευρωπαϊκών, τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο μέλλον. Νομίζω όμως και με τις κατεξοδότησης, τις που αναφέρεται τι θα γίνει στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση μεταρρύθμισης για την ισοδυναμία η οποία προσαρμόζεται σε αυτήν την θέληση εξυγχρονισμού του συστήματος ισοδυναμίας προκειμένου να είναι κατάλληλη για το σκοπό που προσπαθεί να επιτύχει. Εκεί συμφωνώ και συμφωνώ και με το θέμα της διαφάνειας που έθεσε ο εισηγητής. Ε, φαντάζομαι ότι η Επιτροπή μας θα μπορέσει να επεξεργαστεί ε, την συγκεκριμένη έκθεση και να καταλήξει σε ε, απόφαση που θα είναι υπέρ της διαφάνειας. Το θέμα είναι όμως ποια είναι η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρόκειται για διαδικασία πολιτικής διαιτησίας αν ο εισηγητής ε, απέφευγε αυτό το κίνδυνο, τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ε, να ευνοηθεί το σύστημα ισοδυναμιών που υπάρχει αυτή τη στιγμή, επαόριστον ε, μετά από αξιολόγηση σημείο προς σημείο ε, των ε, στοιχείων όλων που πρέπει να αξιολογηθούν. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να ξαναδούμε σε αυτήν την έκθεση. Υπάρχουν στοιχεία πολύ σημαντικά και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θέλουμε βέβαια να καταλήξουμε σε μια διαδικασία που θα είναι προ συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η παράγραφοι 5, 8, 9, 15, 17, 20 και 23 του σχεδίου έκθεσης ε, πρέπει να αναδιατυπωθούν ε, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αν όχι να αναδιατυπωθούν ε, εντελώς. Forgive me. Μόλις το συγγνώμη, αλλά τα βλέπουμε γυαλιά Brexit τα πάντα. Αυτή την προοπτική έχω αυτή τη στιγμή και θέλω να με καθησυχάσει ο εισηγητής ε, γιατί το φοβούμε ε, να μπει το ΣΥΤΙ στη μέση και να τα κάνει άνω κάτω ε, στα ενένια αγορά κάποια στιγμή. Ελπίζω λοιπόν να μην συμβεί αυτό σε καμία περίπτωση. Καταρχά είναι σαφέ ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ρύθμιση. Πώς θα επηρεάσει όμως Εμεί τώρα λέμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα προβεί σε απορρίθμιση, άρα πρέπει να μειωθούν τα πρότυπα. Ή λέμε ότι μπλοκάρουν κάποια νομοθετήματα οι Βρετανοί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό που εννοούμε και πώς θα επηρεάσει δηλαδή η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου τη ρύθμιση σε ό,τι αφορά την ισοδυναμία της είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα και δουλεύει πολύ καλά. Η έκθεση λέει ότι μπορεί να προωθηθεί περισσότερο διεθνή συνεργασία με διεθνεί συμφωνίε που διαπραγματεύεται η Ένωση με τι τρίτε χώρε σε είδο ε, πλαισίου ελεύθερου εμπορίου. Ο εισηγητή είπε στην ομιλία του ότι πιστεύει ότι πρέπει να είναι αμφίδρομο το σύστημα και όχι εμεί να έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα και να περιμένουμε να τα φτάσουν οι άλλοι. Έτσι βλέπω και την ε, ισοδυναμία και εγώ και αυτό θα συνεχίσω να υποστηρίζω. Στην παράγραφο 9 λέει ότι η διαργασία για τη χωρίς ισοδυναμία στερείται ασφάλεια και παρκώς διαφάνεια και χρειάζεται ένα δομημένο και λειτουργικό πλαίσιο. Ναι, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε την αποδυνάμωση και την άσκηση πέσεων. Και στην παράγραφο 10 λέει ότι οι αποφάσει ισοδυναμία και διεθνεί συμφωνίε θα πρέπει να είναι αντικειμενικέ, αναλογικέ, ευαίσθητε σε θέματα και δεν καταλαμβάνονται προ το συμφέρον τη Ένωση και των πολιτών τη και εγώ θα έλεγα και για την προστασία τη νέα αγορά που είναι και προς συμφέρον των πολιτών βέβαια αυτό. Αλλά όπως είναι αυτή τη στιγμή διατύπωση, οι πολίτες θα έχαναν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν κάποιες επιχειρηματικέ δραστηριότητες. Άρα καλύτερα ε, να λάβουμε εδώ υπό κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με το City. Η πράσπιση της εσωτερικής αγοράς νομίζω είναι το σημαντικότερο. Η ισοδυναμία πρέπει να είναι μονόδρομος νομίζω για τα ανώτατα υψηλά πρότυπα που πρέπει εμείς να πετύχουμε και να ζητήσουμε και από τους άλλους μετά να τα φτάσουν. Εσείς μιλήσατε. Κύριε Κόμπερν, σας είπα ότι ξαναπήρατε το λόγο πριν. Όχι, όχι. No. Oh, I... Mr. Coburn, you, you, first you are not using the microphone. Κύριε Κόμπρα, πρώτα απ' όλα δεν έχετε ανοίξει το μικρόφωνο δεύτερον, και δεν σας ακούει κανένας. Δεύτερον, θα μιλήσετε μόνο να σας δώσω εγώ το λόγο. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος, επειδή μιλήσατε όπως είπα και πριν. Συμφωνούμε? Όπως κρίνετε εσείς σκόπιμο, κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριε Σκόμπριν, πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω κάποια σημεία που θεωρώ σημαντικά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που ο εισηγητής υποστηρίζει την ανάγκη βελτίωσης του μηχανισμού ισοδυναμίας. Και σας υπενθυμίζω και τη δήλωση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και συζητήθηκε με την Διευθύνουσα Ομάδα για το Brexit. Υπάρχει συνένεση και είναι καλό που προχωράμε ως κοινοβούλιο λίγο πιο πέρα και επεξεργαζόμαστε τα διάφορα στοιχεία. Θέλω να πω δύο πράγματα. Φυσικά και δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Αν έχουμε μία πρόταση απλή για τις τρίτες χώρες και την αναθεώρηση της ΕΖΑ, έχουμε το πρώτο βήμα της αναθεώρησης του μηχανισμού ισοδυναμίας, άρα δεν ξεκινάμε εκ του μηδενός. Επεξεργάζομαι κι εγώ μια πρόταση για τα CCBs. Δεν ξέρω τι θα κάνει το Κοινοβούλιο ακριβώς με την αρχική πρόταση. Δεν είναι θέμα μόνο συνέπειες μεταξύ Κοινοβουλίου Κομισιών αλλά και ενδοκοινοβουλιακά. Δεύτερον, για να μην έχουμε παρανοήσεις, όχι ότι το θέλει ο αλλά αυτή η έννοια της αμοιβαίας αναγνώρισης στην παράγραφο 5 και οι φίλοι και οι συνομιλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο το έχουν τονίσει και σωστά νομίζω ο κύριος Μπαρνιέ λέει ότι δεν έχουμε κανόνες αμοιβέ αναγνώρισης στην Ένωση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το ισοδύναμο είναι κάτι διαφορετικό. Ισοδυναμία. Υπάρχει το διαβατήριο βέβαια, που είναι η αγορά όμως. Πέραν του διαβατηρίου υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες που μπορεί να επιτρέπουν κάποια επίπεδα πρόσβαση στι αγορές, αλλά αυτό δεν είναι αμοιβαία αναγνώριση. Και μετά έχουμε την ισοδυναμία. Δεν νομίζω ότι και ο εισηγητή λέει κάτι τέτοιο στα άρθρα τη εκθεσή του. Ότι δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε αμοιβαία αναγνώριση. Μιλάμε για ισοδυναμία, η οποία, το λέει και το Συμβούλιο, είναι πάντοτε μονομερής. Άρα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασίες για να υπάρχει ασφάλεια στους συνομιλητές μας. Δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να είναι αυθαίρετη. Τι θα πει αυτό. Θα πει ότι τελικά είναι όμως μονομερής. Και αυτό θα πει ισοδυναμία. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορούσε να αλλάξει. Άρα η πλαισίωση και η δόμηση δεν θα πει ότι δεν είναι και μονομερές. I, is... Αναθεώρηση είναι απαραίτητη. Αλλά θα ήμουν προσεκτικός. Να μην τα λέμε τόσο αρνητικά για το τι ισχύει τώρα. Ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει ασφάλεια ε, δικαίου κτλ. Μα το σύστημα λειτουργεί. Οι Αμερικανοί φίλοι αντίθετα λένε μην τα αλλάξετε όλα. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί και να θεωρηθεί εν του Brexit το σύστημα. Όμως, όχι τόσο ριζικά. Και να μην είμαστε τόσο επικριτικοί σε αυτό, σε αυτό που ισχύει σήμερα. Επίσης είναι σημαντικός ο ρόλος των εθνικών αρχών και για τις κεφαλαίες όπου δεν υπάρχει νέα αποπτία προς το παρόν, λέω. Φυσικά και θέλουμε οι εθνικές αμμύδιες αρχές να εφαρμόζουν τους κανόνες μας με συνέπεια. Γιατί έχουμε και το ενιαίο rulebook ο ρόλος των εθνικών Υποπτικών αρχών είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και της υποπτικής σύγκλησης για να έχουμε μια ομοιόμορφη εφαρμογή. Αυτή είναι η έννοια και είναι σημαντικό να εισαχθεί αυτό το κόνσεπτ λαμβάνοντας υπόψη και τα πρακτικά στοιχεία που τα γνωρίζετε το λεγόμενο empty shell και τα λοιπά και τα λοιπά πώς θα επηρεάσει το υποπτικό πλαίσιο των Brexit. Και ένας από τους λόγους της ισοδυναμίας είναι να αντιμετωπιστεί ακριβώς ε, το ενδεχόμενο να έχουμε κενά και λήψεις. Και σε ό,τι αφορά τη ισοδυναμία και σε ό,τι αφορά το rule book. Αυτά είναι στοιχεία που η διαπραγματευτική ομάδα είμαι βέβαιος θα τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. Α, έχουμε τον κύριο Κόμπερν και μετά την Κομισιόν. Εξεπλάγει από αυτά τα οποία είπε η κυρία Σκοτ Κέιτο. Στην, στην ουσία... System, the project, whatever, which of course she's fully signed up to by the sound of it. Εν πάση περιπτώσει δεν έπρεπε να είναι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκπρόσωπος της χώρας της. Νομίζω ότι δεν επιθυμεί η Αγγλία να τα πάει καλά στις διαπραγματεύσεις αυτές. Το θέμα εδώ είναι το τι πρόγραμμα ετοιμάζεται και το θέμα είναι να πετύχει το πρόγραμμα και όχι να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. Υπάρχει ένας μεγάλος ε, φόβος με το Brexit ε, και μιας και η Αγγλία έχει πάρα πολλά χρήματα και επενδύει και έχουμε και το City στο Λονδίνο και αρκετά άλλα πλέον εκτήματα σημαντικά και γι' αυτό φοβάστε λοιπόν την αναχώρησή σας. Υπάρχουν και άλλες χώρες όμως όπως και η Ουγγαρία, ίσως και η Γαλλία θα θελήσουν να κάνουν ό,τι κάνει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Διαλύεται η Ευρώπη γιατί ενδιαφέρεστε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι ε, στο ε, συμφέρον των λαών. Ε, μου κάνει τρομακτική εντύπωση αυτό το οποίο είπε η Σκοτ Κέιτο. Ξέρετε ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη συνθήκη, εκπροσωπούν ε, των λαούς της Ευρώπης και των λαών της Ευρώπης. Νομίζω ότι δεν είχαν και πάρα πολύ σχέση αυτά τα οποία είπε με το θέμα που συζητάμε. Εγώ πιστεύω ότι η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλή για το συμφέρον των λαών της Ευρώπης και δεν υπάρχει καμία σύγκρουση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωσης και στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. Νομίζω ότι τα συμφέροντα των λαών προστατεύονται όταν έχουμε ισχυρούς χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς και εμείς προσπαθούμε ακριβώς αυτά τα συμφέροντα να υπερασπιστούμε. Σας ευχαριστώ. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρία σημεία δεν λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση όλες τις προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει και για τις νέες εποπτικές αρχές και για το ΕΜΙΡ και τα λοιπά. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα το 2017 και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα δεύτερο σημείο σχετικά με την αμοιβαιότητα. Στην ουσία ή στην πρακτική οι ισοτιμίες δείχνουν ότι μπορούμε να πετύχουμε αρκετά επίπεδα αμοιβαίας αναγνώρισης με ένα ελεγχόμενο τρόπο και δεν είναι σωστό λοιπόν αυτό το οποίο ακούστηκε ότι μόνο μέσα από αμοιβαία συμφωνία μπορεί να πετύχει κανείς τους στόχους αυτούς. Και αυτό απεδείχθηκε στα πλαίσια των συνέχειας που δόθηκε στις αποφάσεις για τη ΜΥΦΕΔ και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ε, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τις ΕΠΑ. Τώρα για την Ελβετία. Η αναφορά είχε σχέση ακριβώς με μια διαπραγμάτευση που δεν είχε ολοκληρωθεί και το θέμα δεν ήταν κάτι το διαφορετικό και γι' αυτό ακριβώς η απόφαση ήταν αυτή που ελήφθη. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και θα μου επιτρέψετε να δώσω κάποιες απαντήσεις. Εγώ ξέρω ποιες είναι οι δυσκολίες τις οποίες έχουμε εμείς σαν Ιρλανδοί σε σχέση με τον Brexit και δεν τις απέκρυψα και θα ήθελα να έχω μια έκθεση η οποία θα τύχει υποστήριξης από την πλειοψηφία και ωφέλιμης για το μέλλον και δεν είναι κάτι το οποίο θέλω εγώ να προτείνω πως για λόγους προσωπικού συμφέροντος γιατί επειδή είπατε ότι επειδή είμαι Ιρλανδός δεν θα μπορούσα να είμαι δίκαιος δεν είναι σωστό σαν παρατήρηση. Υπήρξε επίσης μια παρανόηση της ερωτησής μου στην αρχή όταν ρώτησαν το σύστημά μας είναι το κατάλληλο. Δεν ήταν δήλωση αυτό, ήταν ερωτηματικό. Συνεπώς λοιπόν εγώ δεν προτείνω μια ριζοσπαστική απόκληση από το νομικό πλαίσιο παρά την επιθυμία την συστηματική ορισμένων να παρανοήσουν αυτά τα οποία λέγω. Εγώ ζητώ να υπάρξει μια προσαρμογή έτσι ώστε πρώτον να έχουμε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο, όχι επιμέρους αποφάσεις, δεύτερον οι διαδικασίες να είναι ξεκάθαρες για όλους και για αυτούς οι οποίοι ετούνται αν θέλετε δικαιωμάτων και στο τέλος ο μηχανισμός αναθεώρησης να είναι πιο ξεκάθαρος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να περάσουμε σε ένα σύστημα κοινοβουλευτικού ελέγχου των αποφάσεων που λαμβάνονται. Όχι εμείς να παίρνουμε τις αποφάσεις, αλλά να ελέγχουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Και γι' αυτό θα ήθελα όλες οι τρίτες χώρες, οι σχέσεις τους ε, με εμάς να βοηθηθούν. Τώρα για την αμοιβαία αναγνώριση. Είναι σαφές ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα λεγόμενα δικαιώματα διαβατηρίου, passport rights. Είναι ένα σύστημα το οποίο ανήκει σε μας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθιερωμένο σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές και ισχύει για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν επίσης και τα συστήματα ισοτιμιών. Έχουμε επίση και συστήματα αμοιβαίων αναγνωρίσεων σε πολλούς τομείς όπως στην ασφάλιση, στην αντασφάλιση με τις Ηνωμένε Πολιτείε Έχουμε παραδείγματα εκεί και ισχύει το ότι ε, προσπαθήσαμε στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ να υπάρξει ένα ξεκάθαρο κεφάλαιο για τα χρηματοπιστωτικά. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο προτείνω και στην παράγραφο 5 και δέχομαι κύριε Φερνάντες ότι θα πρέπει να διορθωθεί αν θέλετε η διατύπωσή της, ότι δεν είναι μία απόκληση ριζοσπαστική από τις αρχικές μας θέσεις ή από τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Τώρα για τις εποπτικές αρχές σε σχέση με, τις, με τα MCA. Σε σχέση λοιπόν ε, με τις ε, εθνικές αρχές ε, και πώς μπορούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου να αναγνωριστούν. Εγώ είπα ότι η λήψη αποφάσεων όπως λαμβάνεται ή γίνεται μάλλον σήμερα από τις εθνικές αρχές δεν ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είναι βέβαια πολιτικό το θέμα, το παραδέχομαι αυτό και πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι ε, αναγνωρίζουν την ε, ισορροπία η οποία χαρακτηρίζει την έκθεση. Εγώ δεν θα ήθελα η έκθεση αυτή να θεωρηθεί σαν αντίβαρο στις ε, ε, διαπραγματεύσεις οι οποίες διεξάγονται για τον Brexit την παρούσα φάση. Θα ήθελα όμως να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερος ρόλος του Κοινοβουλίου στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι σήμερα είναι αποδεκτό σημαντικές αποφάσεις για τρίτες χώρες να λαμβάνονται χωρίς τον έλεγχο μας ε, και χωρίς οι διαδικασίες να είναι ξεκάθαρες και νομίζω ότι αν το πετύχουμε αυτό θα έχουμε πετύχει κάτι θετικό και νομίζω ότι και μετά και από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα το πετύχουμε. Συνεπώς λοιπόν ε, μπορούμε να πετύχουμε μια πλειοψηφία η οποία να στηρίξει την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα το χρονοδιάγραμμα. Α, μια στιγμή, μια φράση ακόμα λέει ο εισήγητης. Ζητά συγγνώμη ο κύριος Φόξ, μου έστειλε τις παρατηρήσεις του. Είναι σκιώδης των συντηρητικών και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις παρατηρήσεις του κύριου Φόξ συνεπώς. Δεν μπορούμε εμείς παρά να τις αγνοήσουμε, λέει ο Πρόεδρος, γιατί δεν μας τις έστειλε σε εμά, αλλά θα μας τις δώσετε. Λοιπόν, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 12η μεσημβρινή την επόμενη Πέμπτη, 28 ε, Μαΐου και 18 και 19 η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και τον Σεπτέμβριο θα φτάσουμε στην Ολομέλεια. Λοιπόν, τελειώνουμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε αύριο στις 11. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε.